καταψήφισα τον σημερινό προπολογισμό. Γιατί προτείνει αύξηση στις δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 6,8%. Το να ζητάει τέτοια μεγάλη αύξηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιαδήποτε αύξηση, είναι παράλογο και ε, δείχνει έλλειψη ευαισθησία. Θα απομακρύνει του ψηφοφόρου του Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ένωση. Γιατί η Ευρώπη θα παίρνει, πρέπει να παίρνει περισσότερα χρήματα, ενώ όλε οι δημόσιε υπηρεσίε παίρνουν λιγότερα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνει κήρυγμα στην Ελλάδα, ζητάει από την Ιρλανδία να, μειώσει τους, ε, ε, να αυξήσει του φόρου και από την Ισπανία να προσφύγει στο μηχανισμό διάσωση και αυξήνει τα δικά τη κονδύλια. Είναι υποκριτικό υποστηρίζω τις προσπάθειες του David Cameron να παγώσει τις δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιο κοντά στους ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, από ότι το πολλά από τα μέλη του Σπάταλου Κοινοβουλίου. George Lyon? think left. Grazie. Ευχαριστώ. Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η πολιτική λιτότητα που εφετήθηκε την έξοδο την οικονομική κρίση δεν έδωσε τα αποτελέσματα που ελπίζαμε. Όπω υπογραμμίστηκε από την έκθεση του συναδέλφου Λαδία, μόνο επενδύοντα με πιο επιλεκτικό τρόπο και υποστηρίζοντα το ιδεώδε ενό προπολογισμού ευρωπαϊκού που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση, θα είναι δυνατόν να εξισορροπήσουμε εκ νέου την οικονομία των κρατών μελών Βελτιώνοντα την κατάσταση για του Ευρωπαίους πολίτε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εξέφρασα την ψήφο μου υπέρ της εκθέσεως αυτής. Ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Το καθήκον των Ευρωβουλευτών είναι να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ε, ψηφοφόρων τους. Ε, η εμπιστοσύνη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον ΑΔΙΡ σύμφωνα με το Eurostat, λιγότερο από το 1 τρίτο των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δική μου χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ως ε, ε, απομακρυσμένη και σπάταλη. Αν θέλουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη θα πρέπει να χαλιναγωγήσουμε τα υπερβολ, τις υπερβολικές δαπάνες. Η αύξηση κατά 7 περίπου του υπερπολογισμού, η πρόταση αύξηση αποτελεί ε, προσβολή στους δικούς μου ψηφοφόρους. Θα ήθελα να παγώσει τελείω ο προπολογισμό, αλλά η αύξηση του 3% προτείνει το Συμβούλιο είναι επίση δεκτή. Γιατί εμεί λοιπόν ψηφίσαμε να επανέλθουμε στις μη ρεαλιστικές, ε, ε, στα μη ρεαλιστικά αιτήματα της Κομισιόν. Ε, η Κομισιόν πρόσφατα ζήτησε αύξηση 10 δισεκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό του 2012, το δικό της προπολογισμό. Αυτό είναι εξωφρενικό. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κομισιόν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να σπαταλά τους φόρους των πολιτών μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Λαβία και Βόγκαν για την έξοχη δουλειά που έκαναν για τον προπολογισμό 2013 και συγκεκριμένα θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα Erasmus. Από το 87 πάνω από 2,5 εκατομμύρια φοιτητέ Ευρωπαίοι συμμετείχαν και μπόρεσαν να πάνε στο εξωτερικό για να σπουδάσουν και για να εργαστούν. Ψηφίσαμε κατά των περικοπών του Συμβουλίου, ζητήσαμε αυξήσει για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει μόνο να σώσουμε το έρασμο, θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και, όσο, και ακόμα πιο γενικά να προτείνουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους νέου διότι οι νέοι δεν μπορούν να πληρώνουν το κόστος της κρίσης κυρίως ε, σε μια χρονική στιγμή όπου η ανεργία των νέων ε, πλήττει σχεδόν το 20, φτάνει σχεδόν το 25% στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκέρλινγκ απεχώρησε. Ο κύριος Αντωνιώτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κράσω τα συγχαρητήρια προ εκείνο που έκανε ο κύριος Λαβία για την έκθεση για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό του 2013. Ε, ήταν μεγάλο το βάρος του συνάδελφου διότι η συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαινόταν ότι ήταν απόμακρη και δύσκολο να επιτευχθεί. Παρόλο την περίοδο αυτή της κρίσεως και συνεχών αιτήσεων για περικοπέ στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ο κ. Λαβία με τον κ. Βόγκαν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν μια συνέχεια στον αφορά τι πολιτικέ και τι ε, πρωτοβουλίε που έχουν δρομολογηθεί. Είναι σημαντικό, πιστεύω, το ότι απεθεύθη μια επιβράδυνση των πιλωτικών ε, πρωτοβουλειών όσον αφορά το περιβάλλον και την ενέργεια. Είναι σημάδι καλή δουλειά που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπίζοντα τα προνόμια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω πλήρω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Um, Κύριε Γκέρλινγκ. Είμαι me, Mr. President. Sorry. εγώ, Πρόεδρε δεν είναι δυνατόν με τόσους, ε, με περικοπές στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να αυξήσει κατά 3% τον προβληματισμό του 13 κάτι που ε, υπερβαίνει τον πληθωρισμό το Κοινοβούλιο από την άλλη μεριά προτείνει πάνω από 6% αύξηση οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τις, τις ε, εθνικές δαπάνες 83 δισεκατομμύρια λίρες προσπαθεί να περικόψει η Βρετανική κυβέρνηση ε, δεν υπάρχει λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρεθεί από όλη την πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης. Μια ακόμα φορά το Κοινοβούλιο, θα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την επαφή της με το ε, κοινό μας ε, που πλήττεται από τις περικοπές σε εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια, ένα ακριβό εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά θέλει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, να κόψει τις δαπάνες της. Κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεσή του που αποτελεί μια καλή συμβαστική λύση και πιστεύω ότι ο προπολογισμό 2013 βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινή γνώμη. Ούτω ή άλλω είναι το τελευταίο έτος του επταετού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι τώρα και έτσι τα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι μερικές φορές δεν είναι τόσο ακριβοδίκαια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά ήταν τα σχέδια και προγράμματα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ω εκ εισέρευσαν και πάλι στα κράτη-μέλη τα κονδύλια αυτά. Έχουμε ενισχύσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έτσι ώστε και να αρκέσουν και να ε, χρηματοδοτήσουν την καινοτομία, την δημιουργικότητα. Πρέπει να είμαστε ακριβοδίκαιοι ένας με τον άλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Επιτροπή μου, η Επιτροπή δηλαδή εσωτερική Αγοράς, σημείωσε την ανάγκη που υπάρχει για κόστος για το προσωπικό. Δεν πρέπει να ξεπερνά προεπολογισμός τα όρια. Θα πρέπει να εστιαστούμε επιβιώσιμης ανάπτυξης των υποδομών της πληροφορικής, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω του διαδικτύου θα πρέπει ε, να εφαρμοστούν και οι λύσεις για τη θέτηση των διαφορών εξώδικα κάτι που θα υποστηρίξει την εσωτερική αγορά καταψήφισα την έκθεση διότι πιστεύω ότι διάφοροι τομείς χρειάζονται ξεχωριστή ανάλυση και πρέπει να υποστηρίξουμε το Solvit. Yes. Ε, είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό της ε, ρεαλισμού των μελών ε, η απόφαση πήρα μερικά, ε, μερικά λεπτά πιο πριν όλα τα κράτη-μέλη αναγκάζονται να κάνουν περικοπές στις δαπάνες τους και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση το αρνείται αρνείται όλη αυτή την πραγματικότητα παρόλα το ότι επί 16 χρόνια το Ελληνικό συνέδριο ε, την ε, κατακρίνει. Παρ' όλα αυτά, μια, μεγάλο μεγάλος αριθμός ε, βουλευτών δεν ψήφισαν υπέρ της ε, αύξηση κατά 7% πολύ πάνω από τον, από τον πληθωρισμό. Ε, ο κατάλογος των ψηφοφοριών με όλα τα ονόματα θα αναρτηθεί σε όλα τα φόρα του ίντερνετ για να ξέρουν οι πολίτες τι γίνεται με τα λεφτά τους. Κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση διότι η οικονομική κρίση εξακολουθεί να πλήττει την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν μέτρα λιτότητα Τώρα, περισσότερο από ποτέ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράσει υπεύθυνα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών όταν θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό, ήταν εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2013 και οι δημόσιες δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο συνεπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσει προτεραιότητες και θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες αν αυτό παραστεί αναγκαίο. Θεωρώ ότι ο προπολογισμό είναι ένα σημαντικό μέσο για την πρόθεση της ανάπτυξης και τη συνοχής στην Ευρώπη. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο επί της καινοτομίας και του ανταγωνισμού και να προωθήσουμε με καλύτερο τρόπο τις θετικές εξελίξεις στους τομείς αυτούς. Βασική προτεραιότητα για τη Ρουμανία είναι η εξασφάλιση σωστή χρηματοδότηση για τι πολιτικέ συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντέιβιντ έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ο κύριο Ντέβα. Ο κύριος Ντέβα, συγγνώμη. Δεν είναι αποδεκτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά αύξηση 7% ενώ η δική μου ψηφοφοροί, μου εκλογής πρέπει να ε, σφίξουν την ε, ζώνη τους και να τα βγάλουν πέρα με ό,τι έχουν. Και ε, ε ζήτησα το λόγο για να απαντήσω στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο ε, δείχνει να ρίχνει το φταίξιμο στη, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στι εθνικέ κυβερνήσει για την κατάσταση και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι όταν δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται θα έπρεπε να παρακολουθεί τι δαπάνε στα κράτη-μέλη και υπήρχε ένα όριο στο έλλειμμα 3%. Παρ' όλα αυτά αυτό ξεπεράστηκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτε. το, θυμάστε το 3% και το 60% για το έλλειμμα και το χρέος αντίστοιχα. Ε, έπρεπε να τα επιβάλλει η Κομισιόν. Αυτό δεν έκανε. Δεν φαντάζομαι να θέλετε να πάρετε το λόγο για την έκθεση Berg Κάλφιν. Ωραία, αφού θέλετε να μιλήσετε και γι' αυτό, ξανασηκωθείτε. Άλλο ένα λεπτό. Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 14-20. και Κάλφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή ψήφισα με την ομάδα μου εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που αφορούσαν διεθνείς εξελίξεις διότι δεν πίστευα ότι παρόλο που εμείς αντιμετωπίζουμε δυσκολίες δεν πρέπει να τιμωρήσουμε που εκείνους που είναι σε τόσο κακή οικονομική, ανάπτυ... οικονομική κατάσταση. Και ζούμε στην πολυτέλεια στην Ευρώπη σε σχέση με τον τρόπο που ζουν οι άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο. Και γι' αυτό για τα προγράμματα της φτώχειας και για τα άλλα προγράμματα που έχουμε κάνει περικοπές κυρίως για την Ασία Εκεί διαφοροποίησα τη θέση μου σε σχέση με την ομάδα μου. Διότι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνδέσουμε τη δική μας ευμάρεια με την καλή ποιότητα ζωή των άλλων που ζουν σε πολύ σκληρές συνθήκες και σε περιστάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο καλές όσο αυτές που, στις οποίες ζούμε εμείς. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζανίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο συζητούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο την περίοδο 2014-2020 είναι προβληματικό. Τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν εφορολογικές και οικονομικές περικοπές ε, σε εθνικό επίπεδο για να εξηγιάνουν τα δημοσιονομικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιες περιστάσεις φαίνεται σαν μια οντότητα που μεγαλώνει το οικονομικό βάρος των φορολογουμένων. Γι' αυτό, για να βγούμε πραγματικά από την κρίση και να εγγυηθούμε ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους Ευρωπαίους, θα είναι θεμελιώδος σημασία να υποστηρίξουμε μεγαλύτερες και πιο σημαντικέ επενδύσει στου τομεί τη εκπαίδευση, κατάρτιση και τη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιανακουδάκη. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Μάργαρετ Θάτσερ γιόρτασε τα 87 γενέθλιά της και είμαι σίγουρη ότι θα θέλαμε όλοι μαζί να τη συγχαρούμε. Η κυρία Θάτσερ ε, διαπραγματεύτηκε ε, ε, το Βρετανικό τσέκ το 1994 όταν, όταν δέχτηκε ε, την επιστροφή του 60% της εισφοράς της, ε, της Βρετανίας είχε πει θα προτιμούσα το 100% αλλά ε, πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι και η Βρετανία εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη. Ε, η πρόταση της εξάλληψης ε, της επιστροφής ε, της σύνσφορας στη Βρετανία είναι απαράδεκτη. Και ο κύριος Κάμερον και η κυρία Θάτσερ είχε, είχαν επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα εκείνων των διαπραγματεύσεων που ήταν καλά και για την Ευρώπη και για τη Βρετανία. Γι' αυτό το λόγο η Βρετανία ζητά πάγωμα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι λογικό, δεν καταλαβαίνω πώς η Κομισιόν μπορεί να, ζητά, να συνεχίζει να ζητά αύξηση στο δικό της προπολογισμό ενώ επιβάλλει με μέτρα στα κράτη-μέλη. Ως πρώην επιχειρηματίας γνωρίζω ότι είναι δυνατόν να γίνουν περικοπές σε οποιοδήποτε προϋπολογισμό. Οι πολίτες μας ε, τις αξίζουν αυτές τις περικοπές και η Κομισιόν πρέπει να ακούσει τα αιτήματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε καιρού κρίσεως που ζητούν μείωση τα κάτι μελη των κοινοτικών εισφορών τους, θα πρέπει να δαπανούμε καλύτερο τρόπο θέσιμους πόρους, χρησιμοποιώντας τους για τις πραγματικές προτεραιότητε, ανάπτυξη, απασχόληση, κόβοντας τι δα... σπατάλες και θα πρέπει να ακολουθούμε σωστή προσέγγιση. Θα πρέπει καταργηθεί το σύστημα των μειώσεων ε, του προϋπολογισμού ε, που έχουν και επιστροφής χρημάτων που έχουν προνόμιο κάποια κράτη ε, εναντί άλλων. Η επιστροφή χρημάτων η Βρετανική είναι κάτι απαράδεκτο που αντιστοιχεί στο περίπου 97 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χώρα μου η Ιταλία δεν μπορεί να επιτρέψει την πολυτέλεια αν είναι καθαρός συνεισφορέας και να δίνει περισσότερα από αυτά που εισπράττει. Κυρίως δεν μπορεί να πλέον να το κάνει ούτως ώστε να χρηματοδοτεί αυτούς τους λογαριασμούς τους αναχρονιστικούς. Το 2011 είχε αρνητικό ισολογισμό περίπου 6 δις ευρώ η Ιταλία. Όσον αφορά την Ιταλία και τις πατάλες, να πω ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα, ούτω ώστε γρήγορα να φτάσουμε, ε, να έχουμε μία και μοναδική έδρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ το μεσοπρόθεσμο διευθυντικό πλαίσιο ε, καθορίζει τον ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια έτσι, ε, και είναι επίκαιρο. Όλα τα κράτη-μέλη κάνουν περικοπές ε, σε, στις εθνικές και τοπικές δαπάνες και οι ευρωπαϊκές δαπάνες θα πρέπει να υπόκεινται στου ίδιους περιορισμούς. Έχουμε περιορισμένους πόρους. Το κάθε ευρώ, το κάθε, η κάθε λίρα, ακόμα και το κάθε σλότι θα πρέπει να συνταπανώνται με πολύ προσοχή. Ε, ε, τα ε, ευρωπαϊκά προγράμματα δείχνουν πολλές φορές ελκυστικά αλλά η γραφειοκρατία τα αυξάνει πάρα πολύ τις σπατάλες θα μπορούσαν πάρα πολλά από αυτά να χρηματοδοτηθούν από, τα τοπικά, από τοπικές ή εθνικές πηγές θέλω να αναθεωρηθεί ξανά να ξαναδούμε ξανά πώς μπορούμε να μειώσουμε τις δαπάνες ξεκινώντας από το δικό μας προπολογισμό αλλά κοιτάζοντας και το δικό μας και το προσωπικό και τις κοινωνικές παροχές έτσι ώστε ε, για όσους εργάζονται ε, επιτοπίως να ισχύει το ίδιο σύστημα σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ήθελα ε, ε τομείς όπως ε, επενδύσεις μπορούν να αυξήσουν την απασχόληση να βοηθηθούν περισσότερο. Ο κ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ε, γίνονται σε ένα πλαίσιο κοινωνικό και οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πάρα πολύ προβληματικό και με δυσαρέσκεια πρέπει να σημειώσω ότι η Ένωση θεωρείται πάντα τους πολίτες σαν μια οντότητα που αυξάνει το οικονομικό βάρος του φορολογωμένου ε, περισσότερο έτσι παρά σαν μια πηγή πολύτιμη. Ε, είμαι πεπισμένο ότι αυτό το γεγονό δημιουργείται το γεγονό ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι σε αντίθεση με του εθνικού προπολογισμού. Σε μια ε, εποχή που έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες που δίνονται στην Ένωση από τη συνθήκη της Λισαβόνα, αλλά και έναντι των σημαντικών πολιτικών αποφάσεων που αναλαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπερψήφισα την έκθεση έχοντας επίγνωση ότι χρειαζόταν ένας διοργανικός συμβιβασμός και ένα σαφές μήνυμα προς τους ε, πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοστέλο. Thank you, Chair το πολιετές ε, μοσομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ε, απαραίτητο έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τις ε, στρατηγικές μας, για παράδειγμα την Ευρώπη 2020. Ε, είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε για να δημιουργήσουμε απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να περικοπεί ή ε, να παγώσει, θα πρέπει να μας πούν ποιε στρατηγικές θα πρέπει να καταλήψουμε. Το 25% του, του Ταμείου Συνοχής θα πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό θα επιτρέψει να συγχρηματοδοτήσουμε προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας των νέων η, ε, η Ιρλανδία έχει αναλάβει δέσμευση για αυτό το θέμα για την δική της ε, Προεδρία. Ε, πιστεύω τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα των ιδίων πόρων και θα ήθελα να συμφωνήσουμε επί ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κύριο Στάνοκ, να συγχαρώ τη δημοκρατία της Κύπρου που αντιμετώπισε το ευαίσθητο θέμα των διαπραγματεύσεων ή το ποτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 με άκρα επιδεξιότητα και είναι η πρώτη εμπειρία που είχε σαν Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτή η νησιωτική δημοκρατία. Οι Κύπροι όπως και η Βρετανία αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει το να παίρνει κανείς αξία για τα χρήματα που δίνει ε, τονίζοντα και την ανάγκη που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργό ο Βρετανό, ο κ. Κάμερον, κατέστησε σαφέ ότι σε περίοδου λιτότητα είναι απαραίτητο για το βρετανικό κοινό να ζητείτε μια αύξηση πάνω τον πληθωρισμό ή να σταματήσει η επιστροφή χρημάτων στη Βρετανία. Δοθέντω, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο συνεισφορέα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προειδοποιηθούν ότι είναι έτοιμο να σκίσει το βέτο του Ηνωμένου Βασιλείου αν χρειαστεί και να πάει σε αιτήσια χρηματοδότηση ανάγκη με παγωμένο προπολογισμό. Μπορεί να περικοπεί πολύ λίπο από τον προπολογισμό. Και το να κλείσουμε την έδρα του Κοινοβουλίου του Στρασβούργο είναι καλή αρχή. Χρειάζεται μεταρρύθμιση η ΚΑΠ και χρειάζεται να μειωθούν τα μία ταμεία, κυρίω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ούτω ώστε μόνο η έρευνα και η ανάπτυξη, ιατρική και επιστημονική να υπογραμμιστούν ή μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών. Για την ώρα, το Βρετανικό κοινό πραγματικά πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα και θα μπορούσε να κάνει πολλά ή καλύτερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Ευχαριστώ, κυρία Κυρία έχει το λόγο. Τα τελευταία χρόνια όλοι αντιληφθήκαμε ότι οι εθνικοί προπολογισμοί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη όλων των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να εξηγιάνουν τα οικονομικά τους. Είναι υπέρ ε, του δημοσιονομικού πλαισίου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξεπεράσουμε την κρίση του ευρώ δίδοντας ε, στα κράτη-μέλη ένα δημοσιονομικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια θα διαρθρώσουν τους εθνικούς προπολογισμού του με έναν τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη. Αν αφήσουμε τα ελλείμματα να αυξάνονται ε, θα βάλουμε περισσότερα ακόμα εμπόδια στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ανάπτυξη. Ο κύριο Γιάρο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα από αυτή τη θέση για άλλη μια φορά να απευθύνω έκκληση προ τα κράτη-μέλη για μια ακριβοδίκη συμπεριφορά και αντιμετώπιση. Δεν είναι δυνατόν να φοράνε την ζακέτα, το κουστούμι των Βρυξελών όταν είναι στι Βρυξέλλε και λένε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να αναλάβει περισσότερε δραστηριότητε και να προβάλλει περισσότερα προγράμματα για καινοτομία και παραγωγικότητα και άρα να τι να τις ζητούν να απορροφήσει περισσότερα χρήματα και μετά με το άλλο κουστούμι όταν γίνουν στι πρωτεύουσέ του να διεκδικούν λιγότερη ε, χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εάν θέλουν περισσότερα αποτελέσματα από τι Βρυξέλλε, τότε πρέπει να δίνουν και περισσότερη χρηματοδότηση και τούμπαριν. Γι' αυτό λοιπόν α είμαστε σωστοί και δίκαιοι ο ένα με τον άλλον. Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση των ε, κρατών μελών, φυσικά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Από την άλλη όμω θα πρέπει και να μεριμνήσουμε ώστε τα προγράμματα που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη και την ενεργοποίηση και πάλι τη οικονομική ανάπτυξη να χρηματοδοτούνται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο ο προπολογισμό εφαρμόζεται και από τα νέα κατημέλη όπω και την Πολωνία. Και βλέπουμε σαφώ ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται πραγματικά συμβάλλουν στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και ισοτήμων δυνατοτήτων. Αυτή η έκθεση περιέχει πολλά καλά μηνύματα. Επίσης εμπεριέχει όμως και μια προειδοποίηση κατά των περικοπών. Πιστεύω ότι πρωτοβουλίες τη ε, ε, πράξη ενιαία αγορά πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε χρήματα γι' αυτό. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα πρέπει ενεργά να προωθήσουμε και το επιχειρήν. Θα πρέπει η ενιαία αγορά να ολοκληρωθεί. Χρειάζεται και καλή προστασία των καταναλωτών και γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην αύξηση των δαπανών για αυτό το σκοπό. Διότι δεν αρκούν για αυτό το σκοπό για την ώρα. Ευχαριστώ κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. για το δημοσιογικό πλαίσιο για την περίοδο 14-20 και την αντίστοιχη διαδικασία. Είναι ένα ε, βιώσιμο και σταθερό πλαίσιο που θα μπορεί να δώσει εγγύσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και για υψηλό βιωτικό επίπεδο, καθώς επίσης και την ασφάλεια των πολιτών μας ο προπολογισμό τη Ένωση και κυρίω οι δαπάνε σχετικέ με την πολιτική συνοχή ε, είναι ένα ε, σημαντικό μέσο το οποίο θα, πρέπει να εξακολουθήσουμε, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαθέτουν τα κράτη-μέλη για να ξεπεράσουν την κρίση και να πετύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αν επιθυμούμε μια Ευρώπη ανταγωνιστική, βιώσιμη ε, και χωρίς αποκλεισμούς, θα πρέπει να αφιερώσουμε επαρκή κονδύλια στις πολιτικές συνοχές, τουλάχιστον να τις φέρουμε στο ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Θα πρέπει επίσης να καταργηθεί η μακροοικονομική ρεσιμότητα, γιατί, ε, γιατί αλλιώς θα τιμωρούσαν περιοχές που δεν φταίνε για το προβλήματα της εθνικής οικονομίας. Dank u wel, meneer de voorzitter Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω τρία σχόλια να κάνω όσον αφορά το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, τα ποσά έπρεπε να είναι κάπως χαμηλότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει στα όρια των βασικών της ευθυνών. Ήταν πολύ καλή η πρόταση που έκανε την περασμένη εβδομάδα στον ειδικό τύπο ο πρόεδρος Σούλτς. Όμως διαφωνώ με το σχόλιο του για κεντρική αντιμετώπιση των θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλος τρόπος των χρημάτων είναι να χρησιμοποιούνται τα θετικά ταμεία αποκλειστικά στοχότερες περιοχές των κρατών μελών που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Μετά, οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το ΦΠΑ να χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί ε, κρατικές εισφορές. Αυτό δεν είναι κάτι απόλυτα ευκταίο. Τα κράτη-μέλη σπαταλούν λιγότερα χρήματα, όπως βλέπουμε, ε, σε σχέση με τον προπολογισμό για το 2013 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη-μέλη πρέπει να συλλέγουν τους φόρους, να εισπράττουν τους φόρους. Αυτή είναι δική τους αποκλειστικότητα και έτσι πρέπει να παραμείνει. Είναι δύσκολη η καιρή που περνάμε και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ψηφίσαμε νωρίτερα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, ήταν μια από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες που θα πρέπει, έπρεπε να κάνουμε σαν ευρωβουλευτές. Αφορούσε δεκάδες δισεκατομμύρια ε, κορώνες που ψηφίσαμε. Και όσον αφορά την χρήση των χρημάτων από το 2014 με το 2020, ήταν σημαντικό. Είδαμε ότι υπήρξαν και διαμαρτυρίες στην αίθουσα. Η ομάδα μου επέμεινε ότι θα πρέπει να γίνουν ονομαστικές ψηφοφορίες, να ξέρουν οι πολίτες ποιος ψήφισε υπέρ, πού, πότε όσον αφορά τις δαπάνες αυτές. Γιατί μιλούσαμε για τεράστια ποσά. Δεκάδες εκατομμύρια κορώνες. Και είδαμε λοιπόν το πώς λειτουργεί το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πόσο απόμακρη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες. Και δεν υπάρχει επαρκής λογοδοσία. Και δεν αξίζει, να αντιστοιχεί στην δημοκρατία κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ήμουν παρόν για την πρωινή συζήτηση και μπόρεσα με τα χαράς να παράσχω την υποστήριξή μου στις προτάσεις που υπευλήθησαν. Αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως υπόθηκε πρέπει να φτάσουμε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ε, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Όπως έλεγε ο κ. Βαν θα πρέπει να συνεργαστούμε, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούμε και όλοι οι πρωθυπουργοί θα πρέπει να συνεργαστούν. Το άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Εσείς ο ίδιος είστε επιφορτισμένος για την πρόθεση της μίας έδρας ε, του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Θα μειώσει το κόστος, τα ταξιδιωτικά έξοδα θα μειώσει το κόστος κατά περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ για ένα χρόνο και θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη μείωση. Η κυρία Ζαμπόσκα δεν είναι εδώ. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σταθεροποίηση οικονομίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθούν οι επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο προπολογισμό επίση μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Σε αυτή την συγκυρία θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία που έχουν τα υγιή δημόσια οικονομικά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τι προσπάθειές του για να υποφεληθούν τις ε, δυνατότητες ανάπτυξης, βιώσιμης και μόνιμης ανάπτυξης ε, που έχουν. Και το δημοσιοκό πλαίσιο θα πρέπει να δώσει επαρκή δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να είναι δυνατή τα κράτη-μέλη να υποφεληθούν πλήρω. Η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίε σε ό,τι αφορά την, απορροφ... Ε, απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Και οι στόχοι για την περσινή χρονιά και για το... μέχρι το τέλο φετινή αναθεωρήθηκαν. Χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση όμω για την ε, κοινή αγροτική πολιτική. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουν να μειωθούν οι διαφορές ανάπτυξη που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπάρχουν οι απαντήσεις, υπάρχουν οι λέξεις. Ανάπτυξη, απασχόληση, αντιμετώπιση της κρίσης μέσα στον προπολογισμό, αλλά λύση δεν δίνουν η ίδια πολιτική είναι αυτή που οδήγησε την Ευρώπη στο αδιέξοδο και την κρίση. Όλα αυτά τα οποία, για τα οποία επιμένουν ε, με τις πολιτικές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλείσιμο των ε, θέσεων εργασίας ε, και την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεφύγει από το χάος που έχει η ίδια δημιουργήσει. Τον αντίον είναι ακόμα μεγαλύτερο ο κίνδυνο να βυθιστεί περισσότερο στην κρίση προ όφελο και μόνο του, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση, να προωθήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες που αποτελούν οχυρά απέναντι στην κρίση, να δώσουμε ευκαιρίες στην ανάπτυξη, να διαφυλάξουμε την βιομηχανία, να αναζωογονήσουμε την κοινωνική προστασία και άνωθεν και κάτωθεν και να στηρίξουμε το μισθωτό χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει από την κρίση η Ευρώπη. Για την κρίση αυτή δραστηριοποιούμε εγώ μαζί με τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ένα. Για την έκθεση Νταχάνα παρακαλώ. ως μέσα Σπίτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η επόμενη έκθεση αφορά τις ίδιε πόλει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ καταψήφισα όχι λόγω των λεπτομερών αλλαγών που είχαμε επιφέρει όσον αφορά το ΦΠΑ για τα κράτη-μέλη, αλλά Γνωρίζουμε όλοι ότι όταν μιλάμε για τους πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να παίρνει ένα τσεκ, μια επιταγή κάθε χρόνο από τα κάτι μέλη και μόνο, αλλά θέλει να βάλει τα χέρια η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τσέπες του λαού. Θέλει να επιβάλλει τέλος στους, ε, στα καύσιμα για τα αεροπλάνα, φορολόγηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κλπ. Το βασικό θέμα είναι ότι σε όποια ομάδα και αν ανήκει, αν είσαι υπέρ των ευρωπαϊκών φόρων, αφαιρεί τη σχέση μεταξύ των, ε, ε, των πολιτών και τη ε, πρόσβαση στι τσέπε των λαών. Η, Επίτροπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτό το δικαίωμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει, κάνει προτάσει, παίρνει αποφάσεις και έχει, ε, το... δεν εκλέγεται όμως από κανέναν, αλλά μόνο τις κυβερνήσεις. Οπότε η αρχή της, ή των ιδίων πόρων θα πρέπει να καταργηθεί. Δεν ανήκει ε, πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπαζέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ τη έκθεση, γιατί θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος ιδιών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βήμα πρόοδου. Πιστεύω επίσης ότι οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στον φόρο πιστεύμες αξίες μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος αυτός ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών και το καινούριο σύστημα θα είχε και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα μεγαλύτερη διαφάνεια, ελαστικότητα, ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν με αυτόν τον ε, τρόπο να τύχουν ίσης, ισότιμης μεταχείρισης, ε, ενώ θα, μειωνόντουσαν τα φορολογικά βάρη. Όμως υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε αυτή τη διαδικασία. Η μέθοδος αυτή είναι περίπλοκη για παράδειγμα και η διαδικασία απλοποίησης θα είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνονται οι επεξηγήσει ψήφου. Θα ξαναρχίσει η συνεδρία στι 3 το απόγευμα.